θα θεωρήσω εγκεκριμένα τα ψηφίσματα. Μάλλον θα τα διαβιβάσω αρμοδίω τα όσα εγκρίναμε. Ευχαριστώ πολύ που παραμείνατε πέντε συνάδελφοι. Ευχαριστώ τις υπηρεσίες.